Συνάδελφοι, να προχωρήσουμε γρήγορα. Είμαστε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Θέμα είναι η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Καλωσορίζω θερμότατα τους Επιτρόπους Νάρτσετς και Έτιγκερ και τη Γενική Διευθύντρια κυρία Ράιχερτς. Όπως γνωρίζετε η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο από τον πρόεδρο Γιούγκερ και στην ομιλία του για την κατάσταση για την Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασε για πρώτη φορά την ιδέα για ένα ευρωπαϊκό σώμα αλληλεγγύης το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους μεταξύ 17 και 30 ε, ετών να εργάζονται εθελοντικά και στη χώρα τους και στο ε, εξωτερικό προκειμένου να βοηθήσουν τα πλέον ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Λόγω του ότι δεν υπήρχε έως ε, τώρα σαφής νομική βάση η εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας ε, ε, βασιζόταν, βασίστηκε μέχρι στιγμής ε, σε υπάρχοντα μέσα, όπως το Erasmus Plus και η Ευρώπη για τους πολίτες. Αγαπητοί Επίτροπε, θα ήθελα να σας δώσω τώρα τη λόγο για 7,5 λεπτά και αν καταλαβαίνω σωστά η πρόταση που θα μας παρουσιάσετε πριν από λίγα λεπτά μόλις αποφασίστηκε από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Άρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε οι πρώτοι που θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση αυτής της πρότασης και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από πλευράς Κοινοβουλίου θα διαπραγματευτούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Ξέρω ότι ασκείται πίεση και λέτε ότι ε, θα πρέπει τα πράγματα να προχωρήσουν γρήγορα, όμως εγώ πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και Βεβαίως, όσο περισσότεροι συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευση, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και ο χρόνος που θα διαρκέσει, που θα χρειαστεί για την ε, ολοκλήρωση αυτής της πρωτοβουλίας, για την εφαρμογή της. Ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν και αντικρουόμενες απόψεις και αυτό μπορεί πολλές φορές ε, να αφορά και διαμάχες γύρω από το ποιος έχει την αρμοδιότητα Παρ' όλα αυτά σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και στις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο βεβαίως που είναι και αυτό μια απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει το θέμα. Ε, σας δίνω λοιπόν, κύριε Έτιγκερ, ε, θα ζήσω εσάς πρώτα τον λόγο. 7,5 λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευρωβουλευτές, Κύριε Επίτροπε, κύριε Γενική Διευθύντρια, θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία την πρόταση που αποφασίστηκε σήμερα από την Κομισιόν να δημιουργηθεί, να θεσπιστεί μια αυτόνομη νομική βάση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δώσουμε μια προσφορά, να κάνουμε μια προσφορά στη νέα γενιά της Ευρώπης και να της ε, προσφέρουμε μια σταθερή βάση επί της οποίας θα μπορεί να ε, υλοποιήσει την ε, προθυμία της για εθελοντική προσφορά και συμμετοχή στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Βασιζόμαστε στην πολιτική μας εμπειρία, στην πολιτική εμπειρία μη κυβερνητικών οργανώσεων, κοινοφελών οργανισμών, συνδέσμων νεολαίας, φορέων της ε, εργασίας στον τομέα της νεολαίας και στις τοπικές κοινωνίες. Βασιζόμαστε επίσης και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θελοντών και θέλουμε η διαδικασία αυτή να ε, λάβει και ένα ευρωπαϊκό σήμα διασυνοριακό και να υποστηριχτεί και με τα επαρκή χρηματοδοτικά μέσα. Υπάρχει ένα σχέδιο τριών φάσεων. Η πρώτη φάση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πρόκειται για την αξιοποίηση υπαρχόντων μέσων χρηματοδοτικών για να εξασφαλιστεί η άμεση συμμετοχή ε, νέων ανθρώπων 30.000 ε, αιτήσει έχουμε ήδη λάβει, ιδίως από τις ε, χώρες του Νότου, και προκειμένου να αποφευθεί ε, η, η χρονοτριβή, να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να ξεκινήσουν ε, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Με την πρόταση για τη δημιουργία μιας νομικής βάσης της Κομισιόν, παρουσιάζουμε σε εσά και στο Συμβούλιο το, τη νομική βάση που θα αξιοποιηθεί για, το, για τη δεύτερη φάση, 2018-2020. Για την περίοδο αυτή έχουμε επεξεργαστεί μια νομοθετική πρόταση όπου ε, οι βασικότερες ε, νομικές πτυχές ε, βάσει των οποίων ορίζεται αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η ποιότητά του και μέσω της οποίας ε, θεσπίζεται και μια αυτόνομη χρηματοδοτική βάση πρόκειται για 341 ε, εκατομμύρια ευρώ για τα τρία αυτά χρόνια. 90 για το 2018, 119 για το 2019 και 170 ε, εκατομμύρια για το 2020. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ε, σας προσφέρουμε μια σοβαρή νομική βάση προκειμένου να δημιουργηθεί και να χτιστεί εμπιστοσύνη που την χρειαζόμαστε αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε στη διαδικασία αυτή ε, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τους άλλους ε, οργανισμούς, τους άλλους ε, συλλόγους, προκειμένου από τον Ερυθρό Σταυρό στην Ισπανία μέχρι κάποια εθελοντική οργάνωση σε άλλο σημείο της Ευρώπης, στη Φιλανδία, ε, να μπορέσουν όλοι μαζί να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η τρίτη φάση ε, δεν ε, είναι ένα θέμα που επήγε αυτή τη στιγμή. Πρόκειται να ενταχθεί στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και εκεί θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτική βάση μακροπρόθεσμη για 5-7 χρόνια η οποία όπως και η δεύτερη φάση θα πρέπει να επιτύχει ε, το στόχο να μην αποδυναμώσει υφιστάμενα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα ε, κάτι για το οποίο έχουμε δεσμευτεί ε, και εγώ και η συνάδελφος Ναύρατσετς όπως έγινε και με το, με το Erasmus Plus. Η υψηλή ποιότητα θα εξασφαλιστεί μέσω της δημιουργίας ενός σήματος ποιότητας, του Ευρωπαϊκού Σήματος Αλληλεγγύης και όλοι οι εταίροι μας, όλες οι οργανώσεις, οι σύλλογοι, ακόμα και οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν προσφορές ή θέλουν να κάνουν προσφορές σε νέους ανθρώπους στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ε, τηρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για να λάβουν αυτό το σήμα, προκειμένου να μην γίνει ένα dumping όσο προς την ε, ποιότητα και να εξασφαλίζεται παντού η ευρωπαϊκή ποιότητα τόσο πριν αλλά όσο ε, και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος. Τον Απρίλιο έγινε ένα μεγάλο συνέδριο με εκατοντάδες συμμετέχοντες Και εκεί εκφράστηκαν, και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υπέβαλε με την ευκαιρία εκείνη τις δικές του απαιτήσει και ε, θα προσπαθήσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και στην νομοθετική ε, πρόταση αυτή. Σε, εκείνη την, σε εκείνο το συνέδριο, σε εκείνη τη συνδιάσκεψη παρουσιάσαμε τα βασικά δομικά στοιχεία αυτής της πρότασης τα οποία έτυχαν ε, Τη υποστήριξη των ε, περισσότερων. Ξέρουμε ότι οι κοινοβουλευτικέ διαδικασίε είναι σύνθετε, δεν θέλουμε να ασκήσουμε πίεση. Ωστόσο, θέλω να σα πω ότι θα ήταν πράγματι χρήσιμο αν μπορούσαμε μέχρι το τέλο του χρόνου να καταλήξουμε σε συμφωνία προκειμένου ο προπολογισμο απο από 1η Ιανουαρίου του 2018 να μπορεί να προβλέπει ε, κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και ξέρω ότι το Κοινοβούλιο θα εξετάσει την, ε, τον, το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018, θα το κάνει αυτό η Κομισιόν και εκεί θα υπάρχουν και αυτά τα χρήματα, τα 90 εκατομμύρια περίπου που προβλέπονται για το 2018 και με αυτό θα ξεκινήσει ακριβώς και η δεύτερη φάση που σας περιέγραψα ε, προκειμένου να προχωρήσουμε με αυτή την πρωτοβουλία. Συνολικά η προσφορά μας αυτή ε, δεν αποτελεί ανταγωνιστική, η πρωτοβουλία μας αυτή δεν ε, είναι ανταγωνιστική προς την αγορά εργασίας. Δεν θέλουμε να παρακινήσουμε ε, επιχειρηματίες να χρησιμοποιήσουν φθηνό εργατικό δυναμικό διαγράφοντας ή καταργώντας θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις τους. Πρέπει να πρόκειται, θα πρέπει να πρόκειται πάντοτε για θέσεις οι οποίες δεν αμείβονται γενικά στην, ε, στην αγορά εργασίας. Θέλουμε ε, να ε, δραστηριοποιηθούμε σε θέματα κοινωνικής ένταξης, περιβάλλοντος, προσφύγων, ένταξης των προσφύγων και θέλουμε να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία, μια μεγάλη προσφορά έργων, προγραμμάτων, προκειμένου τα οποία θα πρέπει και να ανταποκρίνονται στις τάσεις και στα ενδιαφέροντα της νεολαίας. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής. Ε, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ένας ε, συμμετέχον στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα μπορεί να αποδεικνύει την ε, αλληλέγγυα στάση του και δραστηριοποίησή του. Θα λαμβάνει λοιπόν κάθε συμμετέχον ε, ένα πιστοποιητικό το οποίο θα εξασφαλίζει και θα επιβεβαιώνει και την διάθεσή του, τη διάθεση προσφοράς του, ε, τη διάθεση της εθελοντικής του προσφοράς ε, κάτι που θα αποδεικνύει στην αγορά εργασίας και την καταλληλότητά του να ε, ασκήσει το επάγγελμά του. Πρόκειται δηλαδή για μια προστιθέμενη αξία για, τη, για τους νέους ανθρώπους ε, που θα τους προσφέρει μεγάλες δυνατότητες η συμμετοχή τους σε αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Ελεγγύης Προσβλέπω λοιπόν σε μια βαθιά και σε βάθος μάλλον συζήτηση τους επόμενους, ε, ε, τις επόμενες εβδομάδες και ευχαριστώ για την προθυμία σας για τη συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Κύριε Ναύρασες. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσω εκεί που ο Επίτροπος Έτιγκερ σταμάτησε. το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα σχέδιο για πτήρη αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα θυμόσαστε ίσως ποια ήταν η ιδέα για το Ευρωπαϊκό αυτό Σώμα που γεννήθηκε σε αντίδραση όσον αφορά το δημοψήφισμα του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διότι, όπως δείχνουν και αναλύσεις, η, η συμπεριφορά όσον αφορά την ψηφοφορία άλλαζε ανάλογα με τις ηλικιακέ ομάδες και το κοινωνικό υπόβαθρο και την εκπαίδευση. Όσο πιο εκπαιδευμένοι ήταν οι άνθρωποι, όσο πιο αστεί και νεότεροι οι ψηφοφόροι, τόσο ήταν υπέρ της Ευρώπης. Η εμπειρία μας στο Εράσμους και το Εράσμους Plus ποια ήταν. Ότι το Εράσμους μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά, μπορεί να αναπτύξει ένα συνέστημα ευρωπαϊκής ταυτότητας, έχει απτά στοιχεία, κινητικότητα των φοιτητών, εθελοντισμό. Ας δώσουμε λοιπόν μια ευκαιρία για εθελοντισμό. Σαν μέσα στα πλαίσια ειδικού σχεδίου, ξεχωριστό νομικό πλαίσιο, περισσότερα χρήματα, εύκολη πρόσβαση, ούτως να συμμετέχουν περισσότεροι νέοι, ούτω ώστε να έχουν εμπειρία τη Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και του ευρωπαϊκού τρόπου να παρέχει κανείς εθελοντικά υπηρεσίε. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τις πρώτες δομές ε, στα πλαίσια του Έρασμους. Δημιουργήσαμε μια θηρίδα στο διαδίκτυο που είναι ένα μοναδικό σημείο επαφής εισόδου όπου μπορούν να υποβάλλονται προσφορές, οι ΜΚΟ μπορούν να στείλουν τις προσφορές τους για εθελοντισμό και υπάρχει και πλευρά της ζήτησης της πύλης αυτής. Είναι νέοι πολίτες ε, μπορούν να καταχωρηθούν και να υποβάλουν αίτηση για εθελοντισμό ή κάποια μαθητεία, αν θέλετε. Περίπου 30.000 νέους είχαμε μέχρι τώρα κυρίως από τα νοτιοευρωπαϊκά κράτη που έχουν δηλώσει συμμετοχή 5.352 ανθρώπους από την Ιταλία 4.470 από την Ισπανία 2.836 από την Πορτογαλία οι πρώτες τρεις χώρες όπου ήδη είναι πολύ δημοφιλές αυτό το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντισμού, είναι αυτές. Υπάρχει ε, αποδοχή των ευρωπαϊκών αξιών εκεί και ταυτόχρονα θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν καλή εμπειρία όσον αφορά την μαθητεία ή τον εθελοντισμό. Γι' αυτό διευρύναμε την έκκληση για αυτό το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα όπως είπε και ο Επίτροπος Έτιγκερ, έχουμε δύο σκέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελληνικής. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον εθελοντισμό, αποτελεί περίπου 80% των δραστηριοτήτων και το τμήμα της απασχόλησης, σκέλης απασχόλησης 20% των δραστηριοτήτων και προπολογισμό. Ακροθυγώς στρέφομαι προς τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ε, είναι EVS ε, συν εκτός από μια άλλη διάσταση. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καλύπτει γεωγραφικά 28 κράτη-μέλη. Ενώ το EVS και το Erasmus καλύπτουν 33 κράτη. Θα υπάρξει ταυτόχρονη ύπαρξη, συνύπαρξη για μη χρονική περίοδος, περίοδο συγγνώμη, για τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Σώμα Αλληλεγγύης θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητε ενώ στις χώρες γειτονίας το EVS θα εξακολουθεί να ζει για κάποια περίοδο. Το Ευρωπαϊκή Θεωρητική Υπηρεσία. Θέλουμε την πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να την κάνουμε πανεύκολη ε, για τα μη κράτη-μέλη μπορούμε να διευρύνουμε ε, το γεωγραφικό πεδίο στις χώρες εκείνες, εκείνες που δεν ανήκουν σε αυτή τη φάση στις δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, οπότε μπορούμε να καλύψουμε τελικά και τις 33 χώρες στο μέλλον. Στην πρώτη φάση όμως Υπάρχει Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής και θα υπάρξει Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα για δραστηριότητες στα πλαίσια των χωρών της πολιτικής γειτονίας. Όλες οι άλλες διαφορές αποτελούν πλεονεκτήματα και μόνο για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διότι όπως προανέφερα η πύλη στο διαδίκτυο θα είναι πιο προσβάσιμη από το πρόσφατο σύστημα της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Εθελοντισμού. Εξακολουθούμε να κρατούμε όλες τις καλές συμπράξεις, εταιρικές σχέσεις, αδειοδοτημένες ΜΚΟ, με τις οποίες συνεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια της περίοδου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού. Θα έχουμε περισσότερα χρήματα και ο μηχανισμός μίας και μόνο θηρίδας για τις αιτήσει καθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εύκολη για τους ετούντες, για τους νέους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν μπορούμε να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό αυτό σώμα και διατηρήσουμε τη λειτουργία του συστήματος όσον αφορά τον εθελοντισμό, θα είναι κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που ήταν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού. Από την άλλη πλευρά, το θέμα της απασχόλησης, η ποιότητα είναι το πιο ευαίσθητο, της μαθητείας και της κατάρτισης. Οπότε, προσδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στη διαφύλαξη όλων των ποιοτικών κριτηρίων που βοηθούν τους νέους να πλησιάσουν μία εμπειρία ποιοτική όσον αφορά τη μαθητεία και την κατάρτιση μέσω των σχετικών προγραμμάτων. Γι' αυτό το πλαίσιο είναι πιο στενό, διότι υπαγρυπνούμε περισσότερο όσον αφορά τα θέματα που άπτονται σε απασχολήσεως. Είναι πιο επικίνδυνος τομέας, διότι έχουμε μικρότερη εμπειρία όσον αφορά την ανάπτυξη των προγραμμάτων μαθητείας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ενώ έχουμε πολλή εμπειρία όσον αφορά την υπηρεσία αλληλεγγύης. Αυτά λοιπόν είχα να πω εντός 7,5 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλά. πολύ Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στους συντηρησίες ξεκινώ σε αυτή τη συζήτηση και έπειτα θα έχουμε ένα δεύτερο ε, γύρο. Ο κύριος Έτιγκερ βέβαια πρέπει να φύγει στις 11. Δεν ξέρω αν υπάρχουν θέματα για τον προπολογισμό που θα μπορούσε ίσως να απαντήσει πρώτα Κυρία Σαμπίνε ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστώ και τους δύο που είστε εδώ σήμερα το πρωί για να μας παρουσιάσετε αυτό το νέο project, που νέο project βέβαια είναι το 20% ουσιαστικά κατά την άποψή μου, γιατί ουσιαστικά ε, παλιά και γνωστά είναι τα 80% του περιεχομένου, πάντως ε, ε, ξέρουμε ότι είναι σημαντικό το θέμα και του εθελοντισμού. Θεωρώ ότι συνολικά είναι καλή αυτή η πρόταση σε ό,τι αφορά μαθητεία, απασχόληση και εθελοντισμό. Είναι καλό να έχουμε ένα νέο εργαλείο ε, για να μπορούμε να αντλούμε κάποια κονδύλια από διάφορα θέσει του προπολογισμού. Ε, αλλά εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά ένα άλλο όνομα δίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα ένα rebranding είναι ε, και όχι κάτι καινούριο. Σίγουρα θέλω να προωθήσουμε την κοινωνική ανταλλαγή και να βελτιώσουμε τα σχετικά με το κοινωνικό θεματολογία. Έρχομαι σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και έχω κάποιες ερωτήσεις ε, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό ε, για την Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία που γινόταν το, η δράση της στην ευρωπαϊκή επικράτεια, τι θα παραμείνει, γιατί ξέρουμε ότι ουσιαστικά θα αφομοιωθεί από αυτό το ευρωπαϊκό σώμα, τι θα γίνει για ε, το, τη δράση που, και το πεδίο που καλύπτεται εκτός Ένωσης και πώς ε, θα οργανωθεί. Δηλαδή, οι οργανωτικές δομές της αθλητικής υπηρεσίας διατηρούνται για το εξωευρωπαϊκό σκέλος ή υπάρχει συνένωση και για τα έξω εδαφικά, αν μπορώ να τα χαρακτηρίσω έτσι, και Βλέποντας ε, τη νομοθετική πρόταση και συγκεκριμένα τις τροπολογίες στο άρθρο 13 ε, για τον κανονισμό του Εράσμους και τα διατεθέμενα οικονομικά μέσα σε ό,τι αφορά την ε, ενήλικη εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, βλέπω ότι υπάρχει κάποια μείωση. Γιατί έχουμε μία μείωση εκεί, 200 εκατομμύρια. Ε, βλέπω να αφαιρούνται δηλαδή κάποια κονδύλια. Ε, Επίση σε κάποιου άλλου τομεί, εντάξει, λογικό το βλέπω σε κάποιου άλλου τομεί. Και έρχομαι σε ένα άλλο σημείο. Στον προπολογισμό έχουμε αύξηση για τα επόμενα χρόνια, ε, αύξηση των κονδυλίων. Γιατί δεν δαπανίσαμε πάρα πολλά χρήματα και χρειάζεται αύξηση, ιδίως για το Εράσμους, το πρώινα το Κομένιουσα αλλά θέλω να ξεκαθαρίσετε κατά πόσον δεν θα πειραχτούν τα χρήματα που πρέπει να διτεθούν για αυτά τα προγράμματα. Είπατε και για το 2018 για το 2019. Αύξηση του προπολογισμού ε, έχει ζητηθεί. Τελικά τι γίνεται, μειώνονται, βλέπουμε, τι θα κάνουμε αυτά τα ε, κονδύλια. Πρόκειται για φρέσκο, για νοπό χρήμα όπως λέμε. Και τι θα γίνει και με το Εράσμους. Τέλος, μάλλον ένα ακόμη ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες ε, για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, κάτι είπατε για το ερασμου 50, 60, 70%, αλλά δεν βγαίνουν και πολλά χρήματα από άλλα κονδύλια για το Εράσμους. Πρέπει να συντομεύετε παρακαλώ. Ναι, ναι. Το θέμα είναι να ωφεληθούν και άλλοι. Στο θέλουμε την αλληλεγγύη, να προωθήσουμε τη δημιουργία αποδομών και υπάρχουν κονδύλια ε, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το σώμα αλληλεγγύης και όχι μόνο ε, αυτά που ενισχύουν μέχρι στιγμή κυρίως το Εράσμους. Δεν πρέπει να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο το Εράσμους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρέπει να είμαι λίγο αυστηρή λόγω του χρόνου. Γι' αυτό παρακαλώ ο καθένα τρία λεπτά. λίγα Κώστα. Ευχαριστώ. Το εκτιμώ ότι έχουμε εδώ δύο επιτρόπου που εκπροσωπούν αυτή τη σημαντική στρατηγική πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Εγώ πρέπει να πω ότι το πνεύμα και η πρόθεση αυτού του σώματος αλληλεγγύης, γιατί λέμε corps και όχι corp στα αγγλικά, γλωσσικής φύσεως η απορία μου. Είναι μια πρωτοβουλία που χαιρετήσαμε θετικά για τους λόγους που παρετέθησαν και αναφέθησαν από την άποψη της πρόθεσης να δώσουμε προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία στην αλληλεγγύη και να δημιουργήσουμε αυτή την εμπειρία για τους νέους αλλά και διάφορες οργανώσεις που ήδη είναι δραστηριοποιημένες ε, έχουν τεθεί τα θέματα του προπολογισμού. Εστερνίζομαι αυτέ τι απόψει. Θέλουμε να μειώσουμε τον χρόνο. Καλή πολλά σημεία. Να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, εδώ μιλάμε για μια νέα πύλη, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν αίτηση και να γραφούν οι νέοι και να είναι πιο εύκολη πρόσβαση για μια εμπειρία που ήταν αυτή που αναφέραμε για την ευρωπαϊκή ταυτότητα αλλά θεωρώ ότι υπάρχει κάποια σύγχυση όσον αφορά το, ήδη, το είδος της δέσμευσης. Εκτός από τον εθελοντισμό αυτό καθεαυτό και τη σχέση συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων που ήδη κινούνται στα πλαίσια της αντιλεγγύης και στον εθελοντισμό και μπορούν να εργαστούν διασυνοριακά, και όσον αφορά τη μαθητεία, το Tennessee, πέρα από αυτό υπάρχει και άλλη πτυχή που αφορά και μόνο το 20% θεωρώ των δράσεων. Και αυτό αφορά τη δουλειά αυτή καθ' αυτή. Οι οργανισμοί δεν είναι μόνο οι μη κερδοσκοπικοί, οι, οι φορείς που ασχολούνται μόνο με τον εθελοντισμό, αλλά και επιχειρήσεις. Κοινωνικές επιχειρήσεις κατανοώ, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημείο που μας απομακρύνει από την αρχική τοποθέτηση, δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι φορείς ε, που κινούνται σε ένα πλαίσιο, ε, ε, στο πλαίσιο εθελοντισμού. Δεύτερη ερώτηση. Όταν είχαμε συμφωνήσει για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, ζητήσαμε από το Κοινοβούλιο στο Erasmus Plus η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού να έχει περισσότερου πόρου, περισσότερε δυνατότητε να μπορεί να προχωρήσει. Και θυμάμαι ότι είχαμε κάνει σημαντική αίτηση, δηλαδή να προωθήσουμε τα κράτη-μέλη, να σπρώξουμε τα κράτη-μέλη να θετήσουν εθνικού νόμου που θα δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να κινηθούν εθελοντικά ε, και να παρέχουν υπηρεσίε είπατε από τις χώρες που έχουν την εθνική νομοθεσία, όχι μόνο από τις χώρες του Νότου. Δεν θα ήθελα εμεί να χαθούμε πολιτικά, να χάσουμε πολιτικά την ευκαιρία να σπρώξουμε ότως ώστε να θεσπιστούν εθνικοί νόμοι μεταθέτως το, το σώμα του Ευρωπαϊκού Σώματος ε, Αλληλεγγύης όχι σε διασυνοριακή πρωτοβουλία, όχι για να πηγαίνουν σε άλλες χώρες ή σε φορείς άλλους, άλλων χωρών, να, να κινηθούν εθελοντικά στη χώρα τους. Εάν γίνει αυτό, είναι παρέκκληση από την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Τέλος, και εγώ ανησυχώ για το εξή ότι οι πόροι τελικά είναι περίπου 197 εκατομμύρια από το και 52 περίπου από όλα τα άλλα προγράμματα. Λοιπόν, είναι σωστό να πούμε ότι 80%, 20% όμως είναι σαφές ότι η προοπτική που ανοίγεται είναι αυτή. Δηλαδή να καλύψουμε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θελοντισμού, να την κάνουν πιο γενική. Οι 28 χώρες σήμερα δεν αντικαθιστούν τις 33, αλλά εδώ τίθεται το άλλο θέμα. Ο Ευρωπαϊκό εθελοντισμό αφορούσε και τι τρίτε χώρε. Είναι εθελοντισμού διεθνού συνεργασία. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με αυτό. Και αν διαρκεί μόνο μέχρι το 2020. Και αν υπάρχει νέα προοπτική μετά το 2020. Και μπορεί όλο αυτό να ξανανοίξει σαν πλαίσιο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διευκρινίσουμε περί τίνο συζητούμε, ποια είναι η νομική φύση ε, αυτής της ε, εμπειρίας που θα είναι εθελοντισμός, αλληλεγγύη, μαθητεία, απασχολησιμότητα ή είναι δουλειά και επιχειρήσει. Ε, αυτό είναι κάτι εντελώ διαφορετικό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σχοντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους επιτρόπους που είχαν την καλοσύνη να μας ενημερώσουν και μάλιστα από πρώτο χέρι, καθώς ορισμένα αποφασίστηκαν μόλις πριν από ό,τι άκουσα. Ε, ομολογώ ότι ε, ε, είχα ετοιμάσει ορισμένα ερωτήματα, αλλά και από τις τοποθετήσεις των επιτρόπων μου δημιουργήθηκαν καινούρια ή ορισμένες διαστάσεις των ερωτημάτων, καθώς αναφέρθηκαν κάποιες πλευρές από τους συναδέλφους. Πιο συγκεκριμένα, αφού θα παρακαλούσα τους επιτρόπους που έχουν τη λίστα μπροστά των πρώτων εθελοντών να μου έδιναν και το στοιχείο για την Ελλάδα για να μπορέσω, αν είναι δυνατόν, να βγάλω το συμπέρασμα που είναι και ερώτημα. Πώς το εξηγούν λοιπόν στις χώρες του Νότου που έχουμε τη μεγαλύτερη ανεργία των νέων κατά την ερμηνεία των επιτρόπων να υπάρχει πιο έντονο το στοιχείο του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης. Πώς το εξηγούν αυτό. Και τι πλατφόρμα του προτείνουν. Δηλαδή, αυτός που αναζητεί εργασία πιο έντονα από άλλες περιοχές, τι του δίνουν. Να εμπεδώσει ή να καλλιεργήσει τα ευρωπαϊκά ιδεώδη όπως την αλληλεγγύη, οφείλω να σας το πω και δεν χρειάζεται για ευνοή τους λόγους, δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στην Κομισιόν όσον αφορά το πώς υλοποιεί την υπόθεση της αλληλεγγύης εν γέννη. Αλλά αυτή είναι μια άλλη γενική κουβέντα. Η ερώτηση είναι αυτή. Πώς τι είναι αυτό που κάνει. Και επομένως διασφαλίζεται ότι αυτό που προτείνεται ως πλατφόρμα με πρώτους συγκινημένους, όπως δίνουν τα στοιχεία, τους άνεργους νέους της ε, νοτιοανατολικής Ευρώπης, πώς διασφαλίζεται ότι δεν θα είναι μια λύση δούριο ύπος, θα έλεγα εγώ, για προβλήματα απασχόλησης, ή ε, και πάω στη δεύτερη ερώτηση για να μην σα κουράζω. Πώ εξασφαλίζετε ότι αυτό το σώμα, αυτά, το, αυτοί οι εθελοντέ δεν θα αξιοποιηθούν από κατασκευαστέ μεγάλων έργων μετά από φυσικέ καταστροφέ, υποκαθιστώντα τι ανάγκε για εργατικό δυναμικό. Και βέβαια το τελευταίο είναι μια ανησυχία. Αυτό δεν το έχω δει, πιθανόν στο νομοθετικό σα ε, εκεί πλαίσιο να τα διευκρινίζετε αυτά τα αισθήματα. Τι, τι ρόλο μπορεί να παίξει ή τι βλέπετε μπορεί να παίξει ε, ένα τέτοιο σώμα σε αυτές που λέμε ειρηνευτικές, ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό. Υπάρχει τέτοιο δέσμευση, υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, υπάρχει τέτοια πρόνοια, συζητείτε. Ε, εν υπάρχει απαγόρευση, υπάρχει ότι δεν θα μετέχουν σε τέτοιες αμφιβόλου εν πάση περιπτώσει σκοπιμότητας αποστολές. Σας ευχαριστώ. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα βασικά που μου δημιουργήθηκαν και από την παρουσίαση. Ευχαριστώ κατά τα άλλα την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ πολύ και από πλευρά μου στους δύο επιτρόπους που μας παρουσίασαν τις βασικές ιδέες και τις δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Γενικά θέλω να πω ότι η βασική ιδέα, δηλαδή η δημιουργία πρόσθετων δυνατοτήτων για νέους ανθρώπους να εργαστούν εθελοντικά, ε, θεωρώ ότι είναι σωστή. Και ο λόγος είναι ότι στόχος είναι πάντοτε να ενισχύεται η ευρωπαϊκή συνείδηση και να δίνονται περισσότερες δυνατότητες στους ε, νέους ανθρώπους της Ευρώπης να αποκτούν νέες εμπειρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις αξιοποιούν ε, με γόνιμο τρόπο ε, ώστε να μπορούν να προσανατολίζονται καλύτερα στην ζωή τους. Ε, βεβαίως υπάρχουν διάφορες σκέψεις ε, για το πώς μπορεί αυτό να οργανωθεί καλύτερα, το one-stop shop, η διαχείριση και η διευκόλυνση ω προς την πρόσβαση και την υποβολή αιτήσεων. Όσον αφορά όμως τη χρηματοδότηση, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι την τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού για την υπηρεσία εθελοντισμού υπήρξε διαβεβαίωση από την Κομισιόν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν χρήματα από το Erasmus Plus. Τελικά αυτό δεν συμβαίνει. Παίρνετε λεφτά από το Erasmus Plus και το λέω ξεκάθαρα. Δεν συμφωνώ. Θεωρώ σωστό να δημιουργηθούν αυτές οι πρόσθετες ε, δυνατότητες αλλά όχι εις βάρος του Erasmus Plus. Αν θέλετε ε, και έχετε την καλή, την καλή αυτή βούληση να δημιουργηθεί μια νέα πρωτοβουλία, τότε ναι να το κάνετε, αλλά όχι εις βάρος των προγραμμάτων όπως το Erasmus+. Πρέπει να βρεθούν νέα χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο κριτικής μου και θα ήθελα να σας καλέσω να υποβάλλετε νέα πρόταση, διότι άλλα μας είχατε υποσχεθεί, εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ την πρόταση έτσι όπως την έχετε υποβάλει τώρα. Δεύτερο ερώτημα, που αφορά την ποιότητα. Εμείς θα χαιρετίζαμε αν οι ομάδες εθελοντών μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτόνομα προγράμματα. Αυτό όμως δεν εμφανίζεται στην πρόταση ή τουλάχιστον όχι ρητός. Και θα ήθελα να μου πείτε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να προωθηθούν και να ενισχυθούν δηλαδή αυτόνομες πρωτοβουλίες των ίδιων των οργανώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Από τους συντονιστές δεν έχει ζητήσει κάποιο το λόγο. Γι' αυτό θα ήθελα να δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Έτιγκερ για να μα μιλήσει για τα ζητήματα του προπολογισμού ε, για να μπορέσει και να αποχωρήσει. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, τα κονδύλια για την εθελοντική εργασία, στο βαθμό που επενδύθηκαν για πολίτες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 28 και τα ενισχύουμε. Με αυτόν τον τρόπο τα βασικά προγράμματα του Εράσμους δεν πειράζονται καθόλου. Αντίθετα, ενισχύουμε, εξυψώνουμε την ποιότητα, διευρύνουμε τις δυνατότητες για εργασία στον τομέα της νεολαίας, κάτω από αυτή τη νέα έννοια του σώματος αλληλεγγύης με στόχο να αποτυπωθεί η αλληλεγγύη ως αξία από μόνη της, ως αυταξία λαμβάνοντας βεβαίως χρηματοδότηση ε, και από υφιστάμενα προγράμματα αλλά και με νέα χρήματα. Να το ξαναπώ. Το βασικό, το κλασικό έργο του Erasmus Plus δεν πλήττεται από αυτό το νέο σώμα. Παίρνουμε χρήματα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εργασία και την Κοινωνική Κοινοτομία. 10 εκατομμύρια δεν είναι λίγα για, για την τριετία. Παίρνουμε χρήματα 35 εκατομμύρια συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την τριετία και νέα χρήματα 86,5 εκατομμύρια. Άρα, στοχευμένα για νέους ανθρώπους δημιουργείται μια νέα προοπτική ώστε αυτοί να μπορούν να εργαστούν για ε, κάποιες εβδομάδες ή κάποιους μήνες ε, σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε ευρωπαϊκά project. Συνολικά λοιπόν πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ λαμβάνονται από άλλα προγράμματα αλλά και από καινούργια χρήματα. θέσατε το ερώτημα τι σημαίνει αυτό για ε, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντών και τι θα μείνει σε εκείνη την υπηρεσία. Η λήψη, η αξιοποίηση των ε, χρημάτων για τους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, τα χρήματα, 98 εκατομμύρια ευρώ. 80% δηλαδή ε, των, χρημάτων. 20% ε, κατευθύνονταν σε χώρες εταίρους με τις οποίες θέλουμε να συνεχίσουμε τα project. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό οργανωτικά, αυτό εναπόκειται στους ειδικού. Ε, και θα ήθελα και με τον Πίτροπο Ναύρατσετς να διοργανώσουμε ενδεχομένως και μια διαβούλευση με εμπειρογνώμονες. Το αν θα μπορέσει η δραστηριοποίηση αυτού του σώματος αλληλεγγύης στην περίοδο μετά το 2020 σε γειτονικέ χώρες, αυτό δεν ε, αποκλείεται αυτή τη στιγμή. Να δούμε όμως, μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της πρωτοβουλίας αυτής, μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σώμα αλληλεγγύης και σε χώρες που αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται να αποτελούν πεδίο δράσης αυτού του σώματος. Και στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορεί να υπάρξει και σχετική πρόβλεψη. Γι' αυτό και μιλήσα για τρεις φάσεις. Ε, μιλάμε για την, την πρώτη φάση, την φετινή, δεύτερη φάση 2018-2020, τρίτη φάση μετά το 2020, προκειμένου να μπορέσουμε να οργανώσουμε και χρηματοδοτικά αλλά και τεχνικά ε, όλες αυτές τις δυνατότητες και τη συμπερίληψη τρίτων χωρών γειτονικών. Περιμένουμε με αγωνία τις εκλογές στη Βρετανία και θέλω να σας πω ότι για το σχέδιο προπολογισμού του 2018 η ενδιάμεση ε, αναθεώρηση θεωρήθηκε εγκεκριμένη. Όπως ε, αποφασίστηκε και στο Συμβούλιο θα πρέπει όμως τότε, ε, όπως και τότε μάλλον στην ενδιάμεση αναθεώρηση, ε, μέσα σε ένα μήνα να προχωρήσουμε γρήγορα ε, για να γίνουν οι αλλαγές. Εκεί προβλέπονται 50 εκατομμύρια και στο σχέδιο προπολισμού του 2018 θεωρούμε δεδομένο ότι το, το μπλοκάρισμα που έχει δημιουργηθεί θα αρθεί μετά τις εκλογές του, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν όχι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά αυτά τα 50 εκατομμύρια ε, θα κατευθυνθούν σε, στους δικούς σας τομείς αρμοδιότητας, στο Erasmus Plus. Για, το κριτικό, για, την, ε, για το σημείο κριτικής που ασχήθηκε, για το αν μπορεί κανείς να ε, εμπιστεύεται την Κομισιόν, πρέπει να σας πω ότι εμείς σας παρακαλούμε να μας εμπιστεύετε. Να μας εμπιστεύεστε. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας καλέσω τα επόμενα τρία χρόνια να συμμετάσχετε ενεργά στον διάλογο για να μπορέσουμε να κάνουμε και έναν απολογισμό αν η προσέγγιση που προτείνουμε σήμερα ε, ήταν η σωστή. Δεν υπάρχει ποσόστοση σε κράτο τα Στα ταμεία συνοχή, τα κονδύλια κατευθύνονται με τη μορφή ποσοστώσεων. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που ενδεχομένως να εκφράσουν ε, το ενδιαφέρον τους. Αν τώρα ε, ε, σε, σε σύγκριση με το μέσο όρο είναι πενταπλάσιοι οι νέοι Έλληνες που θα εκφράσουν το ενδιαφέρον του για αυτό το σώμα αλληλεγγύης, αυτό είναι καταπληκτικό. Γιατί αυτό είναι και προς το συμφέρον της ε, εργασία στον τομέα της νεολαίας. Ακριβώς εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα είναι φυσικό να υπάρχει μεγαλύτερη απήχηση. Δεν υπάρχει ποσόστοση, αντίθετα Καθώς θα εκφράζεται το ενδιαφέρον, θα χρηματοδοτούνται ε, διάφορες δράσεις, διάφορα project και αν ε, ε, είναι ε, περισσότεροι οι Ισπανοί, οι Έλληνες και οι Ιταλοί, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό και θα το χαιρέτιζα. Η Πρόεδρος. Μια ερώτηση πριν φύγετε. 50 επιπλέον εκατομμύρια για το 2017 για το Erasmus Plus και έχουμε άλλα 50 εκατομμύρια που παραμένουν, ελπίζουμε, για το πολιετές δημοσιομικό. Αυτά τα 85 και εκατομμύρια που, που προέρχονται, που είπατε, αυτό το νοπό χρήμα, είναι από τα 100 εκατομμύρια ή όχι, η απάντηση. Global Margin for Commitments για το 2018. Από εκεί προέρχονται, από το 1α, αυτή την κατηγορία. Δηλαδή δεν είχαν διατεθεί ένα συγκεκριμένο στόχο αυτά τα κονδύλια μέχρι τώρα. Και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να επιστραφούν μετά το κλείσιμο λογαριασμών πίσω στα κράτη-μέλη. Και αυτά θα τα καθορίσουμε βέβαια καλύτερα την επόμενη εβδομάδα. Άρα, λέει η Πρόεδρο, αυτά τα πρόστα κονδύλια που λοιπόν, θα πίνει στο Εράσμο για το 2017-2018 κτλ. Ε, μάλλον δεν ε, θα πάνε στο σώμα αλληλεγγύη. Παραμένουν για το ε, υπόλοιπο του προγράμματος Erasmus+. Ναι, αυτός ήταν ο στόχος μας, ε, λέει ο κ. Σέτιγκερ. Το είπα και είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ επιτυχημένη η ιστορία. Να σε ξέρεις τώρα το Erasmus+. Ε, ε, και σίγουρα δεν θα πρέπει να επιβαρύνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στο Erasmus Plus. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλουμε να διατηρήσουμε έτσι τον προϋπολογισμό μας ε, και θα δούμε κατά πόσον μπορούμε και στο μέλλον να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να το αποδυναμώσουμε. Ευχαριστώ. Σας αποχαιρετούμε, χαιρετίστε και τους συναδέλφους από τον προϋπολογισμό. Σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσίαση. Και τώρα περνώ στον Επίτροπο Ναύρατσης, γιατί πραγματικά υπήρχαν και άλλα ερωτήματα. Παρακαλώ, έχετε εσείς τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προβώ σε κάποια συμπληρωματικά σχόλια περί σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Θεωρητικής Υπηρεσίας και Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η βελτιωμένη έκδοση της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Αλληλεγγύης διότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, Αθελοντισμού είναι πολύ δημοφιλές πρόγραμμα, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν ήταν επιτυχέστατο. Σε 20 χρόνια φτάσαμε 100.000 συμμετέχοντες σε μία 20 ετία. Τώρα 100.000 και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το 2020 άλλους 100.000. Με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, σε ένα χρόνο ή λιγότερο από ένα χρόνο, έχουμε 30.000 αιτήσει καταχωρηθήσεις. Μέχρι τώρα είχαμε 108 προσφορές για τοποθετήσεις. Κάποιες από αυτές έχουν υλοποιηθεί, έχουν γίνει τα, οι κατάλληλες τοποθετήσεις αν διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό το Ευρωπαϊκό Σώμα μπορεί να είναι πολύ πιο επιτυχές από την Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία. Όμως, κατάμε, κατάμε κάποια χρηματοδότηση από το Erasmus Plus για εθελοντικές υπηρεσίες σε γειτονικέ χώρες. Έχουμε 90 εκατομμύρια ευρώ ακόμα για δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία στο μέλλον. Αυτά είναι συμπροματικά χρήματα για θελοντικέ δραστηριότητε. Έχουμε τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη, συν 90 εκατομμύρια στο Erasmus Plus για δραστηριότητε Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία στο μέλλον. Και όπως προανέφερα στην προηγούμενη παρέμβασή μου, μπορούμε να διευρύνουμε τη γεωγραφική κάλυψη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης βάσει διμερών συμφωνιών που θα συναυτούν στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να υπογράψει διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες για να, εισαχθεί, εισαχθούν δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη σε αυτέ τι χώρε μέσω διεσυνορικών δραστηριοτήτων. Άρα μπορούμε να επεκτείνουμε την κάλυψη μέσω των δραστηριοτήτων. Η ΜΚΟ είναι ένα πολύ δραστήριο τμήμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέχρι τώρα. Είχαμε 112 οργανισμούς που ήρθαν σε επαφή με συμμετέχοντες, δραστηριοποιούνται, δεν εμφανίστηκαν απλώς στον ορίζοντα, προσπαθούν να βρουν συμμετέχοντες και προσλαμβάνουν συμμετέχοντες. Ε, οι περισσότεροι βέβαια για εθελοντικές δραστηριότητε. Αλλά υπάρχουν και παραδείγματα για απασχόληση, για μαθητεία. Για τέτοιες δραστηριότητε της ΜΚΟ μπορεί να έχετε δυνατότητες για μαθητεία, όχι μόνο για θελοντισμό. Έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα από μικρή χρονική περίοδο και μένεται μέχρι μακρότερη περίοδο για μαθητεία. Η μικρότερη περίοδος μαθητείας είναι δίμηνο. 12 μήνες είναι μεγαλύτερη περίοδος. Στον εθελοντισμό είναι δύο εβδομάδες, η μικρότερη περίοδος και η μεγαλύτερη περίοδος είναι 12 μήνο. Υπάρχει σαφέστατη διάκριση μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Θεωρητική Υπηρεσία και του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη, του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη, είναι βελτιωμένη εκδοχή τη Ευρωπαϊκή Θεωρητική Υπηρεσία. Και θέλουμε να διατηρήσουμε τη χρηματοδότηση σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Σε αφορά την Ελλάδα, μέχρι τώρα είχαμε 1.204 ετούντες από την Ελλάδα, αρκετά καλός αριθμός, 1.204 είναι ο 8 σε μέγεθο αριθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, Ο υψηλό αριθμός ετούντων από τις νοτιοευρωπαϊκέ χώρες μέλη με υψηλό επίπεδο ανεργία των νέων δείχνει το γεγονός ότι αυτοί οι νέοι άνθρωποι όχι μόνο ενδιαφέρονται για την ελληνική και τις θεθελοντικέ δραστηριότητε, αλλά θέλουν να συμμετάσχουν στι δραστηριότητε αγορά εργασία και σε αυτέ επίσης. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μέτρα διαφύλαξης ποιοτικά για να αποκλείσουμε την απογοήτευση αυτών των νέων. Η έλλειψη απασ... Μάλλον θα δίνουμε πιστοποιητικά στον αφορά το τμήμα απασχόλησης του, του Σώματος Αλληλεγγύης και εκείνοι που έχουν προστεί τη μαθητεία και την κατάρτιση θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα πιστοποιητικά στην αγορά εργασίας και ελπίζω να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να βρούνε καλή δουλειά ε, πιο εύκολα. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Τέσσερις ομιλητές έχουμε και θέλω να κλείσω τώρα τον κατάλογο. Ε, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που ακούω εδώ ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από πόρους που δεν θα επιβαρύνουν το, τις δραστηριότητες εθελοντισμού. Χαίρομαι που η πίτροπος είπε ο τελικός σκοπός θα πρέπει να είναι μια βελτίωση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας που υπάρχει τώρα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ή να αφήσουμε εκτός αυτή την υπηρεσία. Δεν πρέπει να απογοητεύσουμε τους νέους οι οποίοι ήδη έχουν ε, καταχωρηθεί να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να απογοητεύσουμε και εκείνους οι οποίοι οικοδομούν την Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία εδώ και 20 χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κάτι κακό, διότι κινήθηκαν σε άλλα πλαίσια και εργάστηκαν οι πάλες συνθήκε. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Θελοντική Υπηρεσία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να κινηθούν παράλληλα, χέρι με χέρι. Διότι ε, θα έχουμε το Σώμα Αλληλεγγύης και την εθελοντική υπηρεσία. Εάν καταργηθεί η Ευρωπαϊκή θελοντική Υπηρεσία θα είναι κακό. Συμφωνώ, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηριχθεί, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υποστηρίξουμε εξίσου και την Ευρωπαϊκή θελοντική Υπηρεσία. Για το κομμάτι εκείνο στο οποίο κινείται. Λοιπόν, θα μπορούσαμε επίση να αλλάξουμε κάπου τον τίτλο για να το καλύψουμε αυτό. Ο κύριος Λόκιγκαρτ ε, ή δεν είναι εδώ ή έφυγε, δεν ξέρω. Ο κύριος ε, Μόργαν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για τι ε, παρουσιάσει. Το, έχω τρει ερωτήσει σύντομες στο χρόνο που έχω θέσει. Πρώτη ερώτηση. Αν κάνω σωστά του υπολογισμού, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Επίτροπο Έτιγκερ, τα δύο τρίτα σε αυτή τη φάση από τη χρηματοδότηση την τριετή από το πρόγραμμα προέρχονται από το Erasmus Plus. Αυτό είναι αυτό που διαπιστώνω. Προφανώς, πώς να το πω, οι ανησυχίες έχουν σημειωθεί. Ε, υπήρξαν και κάποιες χρήσεις αυτών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Εθελοντική Υπηρεσία με τη χρηματοδότηση που πήραμε από το Erasmus Plus από τον τομέα της νεότητας. Αν θυμάμαι σωστά λοιπόν. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι είναι λίγοι πόροι σε σχέση με τις σημαντικούς στόχους, δηλαδή συγκεκριμένη νομική βάση που θέλουμε να δώσουμε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, χρειάζονται οικονομικοί πόροι επαρκής. Δηλαδή αναβάλουμε κατά τριετία το πρόβλημα ουσιαστικά. Πρέπει να πω ότι περίμενα ειλικρινά κάτι περισσότερο. Δεύτερη ερώτηση που θεωρώ που είναι πάλι σημαντικό, σημαντικό σημείο. Απευθύνομαι προς εσάς κύριε Επίτροπε Ναύρασίτς. εσεί είπατε ότι υπάρχουν δύο σκέλη, το Ευρωπαϊκό Σώμα και τη θελοντική υπηρεσία ότι θα συμβιώσουν για μια κάποια χρονική περίοδο. Ε, γιατί, ρωτώ, διότι η εντύπωση που έχω είναι ότι η απάντηση που δώσατε τελευταία είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος, κινδυνεύει το σώμα του εθελοντισμού να μην επιτρέψει πρακτικά να προχωρήσει ο άλλος φορέας. Και μετά πώς βλέπετε εσείς το θέμα της επιλογής, διότι επιμείνατε επί απλούστευσης ε, της επαφής ζήτησης προσφοράς και των προγραμμάτων που υλοποιούνται. Thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον Επίτροπο για απαντήσει. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να βελτιώσουμε την ιδιωτική υπηρεσία. Νομίζω ότι εκείνου από εμά που έχουμε εμπλακεί σε αυτό επί σειρά ετών Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι αναγκαίο σαν βελτίωση. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη είναι μια καλή τέτοια λύση. Καλό τρόπο. Δεν θα μπω σε θέματα οικονομικά. Ο κύριο Έτιγκερ ήδη απάντησε μερικά από τα ερωτήματα. Έχω μια ερώτηση όμω όσον αφορά το θέμα το άλλο. Γι' αυτό που φαίνεται ότι είναι κενό μεταξύ Νοτιοευρωπαίων και Βόρειοευρωπαίων. Την νεολαία αυτών των χωρών όσον αφορά τη συμμετοχή. Λοιπόν, αν ρίξουμε μια ματιά και δούμε τους νέους από τις βόρειες χώρες, ε, ε πώς θα, απευθυνθείτε προς τους νέους της Βόρειας Ευρώπης, ούτως ώστε και αυτοί να συμμετάσχουν. Μιλώντας για αλληλεγγύη, νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικό να ανακαλύψουμε πώς να συμμετάσχουν και οι νέοι από τη Βόρεια Ευρώπη. Οι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα σημείο όπου πρόκειται περί νοτιοευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων που υλοποιούνται. Ευχαριστώ. Μιχαήλ Γκατρούπελ και πάλι. Ναι, για τον προπολογισμό σύντομα να με επιτρέπετε, ξαναείπατε και τέλος πάντων υπέ, υποσχεθήκατε ότι ε, δεν θα αφαιρέσετε κονδύλια του Εράσμους που δεν προορίζονται για θελοντικές δραστηριότητες ε, και είπατε και για τα επόμενα 50 εκατομμύρια. Όμως ε, στην παρουσίαση για την αρχική σας πρόταση, τα 341 αυτά που είπατε, τελικά τα χρήματα που κινητοποιούνται ε, τα πολύ λίγα, πολύ λίγα πηγαίνουν ε, σε αυτό το, το πρόγραμμα. Το θέμα είναι η πολιτική πρόταση και το πολιτικό νήμα που προσφέρουμε ότι τελικά πολύ λιγότερα είναι τα καινούρια χρήματα που συνεισφέρεται σε αυτό το νέο πρόγραμμα. Καλό είναι αυτό που είπατε, δεν θα πάρετε χρήματα από το Erasmus+, απλά εφόσον αυτά δεν προορίζονταν για εθελοντικές δραστηριότητες, αλλά τελικά σε σχέση με αυτό το αρχικό ποσό που ακούγεται, τα 341 εκατομμύρια, αυτό που είναι καινούριο είναι πολύ μικρότερο. Κύριε Νάβατζετς, για να κάνετε τις καταληκτικές σας ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να κάνω άλλη μια απόπειρα διαφοροποίηση τη Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Υπηρεσία με το Ευρωπαϊκό Εθελοντικό Σώμα. Διότι αυτό είναι ο πυρήνα τη νέα έννοια ότι χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση όσο υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Το αισιόδοξο σενάριο ποιο είναι. Ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη υπάρχει συμπληρωματικότητα, γεωγραφική συμπληρωματικότητα, και στο μέλλον θα υπάρξει σύγκληση. Αν υπάρξει επαρκές επίπεδο διμερών συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλων κρατών μελών που πληρούν όλα τα κριτήρια γεωγραφικής κάλυψης, τότε μπορούμε το καλάθι αυτό της Ευρωπαϊκής Στατικής Υπηρεσίας να μπει εντός του Ευρωπαϊκού Σώματος Ελληνικής. Έχουμε εκεί τους πόρους από το Erasmus Plus μαζί με τους εθνικούς φορείς όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στατική Υπηρεσία και την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Σώμα Αλληλεγγύης θα υλοποιηθεί μέσω των εθνικών φορέων. Άρα υπάρχει ένας φυσικός τρόπος συγκλήσεως μεταξύ των δύο αυτών προγραμμάτων και στο μέλλον αυτό θα συμβεί. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση όσον αφορά τις συντονισμένες δραστηριότητε. Σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοιτάξτε, είτε σε όλε τι Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Υπηρεσία είτε το Ευρωπαϊκό Σώμα του Αλληλεγγύη, που θα τα χειριζόμαστε εμεί και εθνικοί φορεί του προγράμματο Εράσμου. Πώ να γίνει δημοφιλέ το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη στη Βόρεια Ευρώπη. Εν μέρει από εσά εξαρτάται επίσης. Αν το προωθήσετε καλά θα είναι δημοφιλές. Όμως μπορώ να σας πω ότι βόρειοευρωπαϊκά βόρειο-ευρωπαϊκά κράτη-μέλη τα πηγαίνουν αρκετά καλά. Ολλανδία που είναι Βόρεια Ελλάδα, Σουηδία καλά τα πάει. Ακόμα και οι Φινλανδοί είναι πιο δραστήριοι από τους Δανούς. Αρκετά εκπληκτικό αυτό. Και οι Βρετανοί είναι αρκετά δραστήριοι. Είναι στο πάνω, στο άνω τέταρτο αν θέλετε. Όσον αφορά το πάνω, στο ανώτερο 25% των ετούντων ειδοπαϊκών σωμαλιλεγγύης πρέπει να βάλουμε μεγάλη πολύ ενέργεια στην προώθηση και διαφήμιση για να ζωγονίσουμε το συνέστημα αλληλεγγύης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να βασιστούμε στα επιτεύγματα του Erasmus Plus, αλλά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Θα πρέπει να εξηγήσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό ενθαρρύνουμε και τους εθνικούς φορείς να κάνουν εκστρατείες ενημέρωσης και διαφήμισης στα κράτη-μέλη και ελπίζω ότι αυτό θα γίνει θετικά αποδεκτό από τους κατοίκους αυτών των χωρών. Για την κυρία Τρούπελ, ναι. Θα θέλαμε να αρπάξουμε όλες τις ευκαιρίες που προέρχονται από όλα τα σχετικά ταμεία Life, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διότι ήδη εκεί υπάρχουν πολύ παρόμοια προγράμματα που ίσως δεν βασίζονται επιθελοντισμού, αλλά επί των ιδίων θεμάτων ε, και θα θέλαμε να ε, εκμεταλλευτούμε όλες τις συνέργειες που έχουν σε αυτά τα προγράμματα. Χρησιμοποιήσουμε όλους τους πόρους από αυτά τα ταμεία επίσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτρο Πενάβρατσες. Χαίρομαι που ήσασταν σήμερα εδώ και μας παρουσιάσατε την πρόταση της Κομισιόν. Επίσημα δεν την έχουμε λάβει ακόμη γραπτός, όπως φαντάζεστε όμως θα την εξετάσουμε όταν τη λάβουμε με μεγάλη προσοχή και βεβαίως θα υποβάλουμε και τροπολογίες κατά τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία. Νομίζω ότι φαντάζομαι δηλαδή ότι στην διάρκεια της διαδικασίας αυτής θα, υπάρχουν, θα υπάρξουν ευκαιρίες να συζητήσουμε με τις υπηρεσίες κομισιών και είναι ε, δεδομένο βεβαίως ότι η συνεργασία μας είναι πάντοτε καλή και θεωρώ δεδομένο ότι ε, η διαδικασία αυτή των συζητήσεων θα φωτίσει διάφορες πλευρές, ε, θα δώσει απάντηση σε ερωτήματα που θα θέσουμε εμείς ως Κοινοβούλιο. Θα συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση η συζήτηση και εδώ στην Επιτροπή, αλλά και μέσα εσάς κύριε Επίτροπε. Και ελπίζω στο τέλος της διαδικασίας αυτής να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα καλό σώμα αλληλεγγύης, το οποίο θα ανταποκρίνεται και σε όλα τα κριτήρια και τις απαιτήσει που αποτυπώθηκαν και στο δικό μας ε, ψήφισμα. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση που βρεθήκατε σήμερα εδώ μαζί μας, ε, που απαντήσατε στα ερωτήματά μας. Θα συνεχιστεί το έργο και ελπίζω, όπως είπα, να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της συνεδρίασής μας. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα γίνει 21 Ιουνίου. από τις 9 έως τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 ε, και το πρωί της 22ης Ιουνίου. Ευχαριστώ τους ε, διερμηνείς για το έργο τους και θα ήθελα να παρακολουθήσω τους συντονιστές να μείνουν στην αίθουσα, όλοι οι άλλοι όμως να αποχωρήσουν. Ευχαριστώ πολύ.